Dear colleagues. Ε, παρακαλώ πολύ καθίστε έτσι ώστε να μπορούμε να ξεκινήσουμε την κοινή συνεδρίαση. Καταρχήν ε, σας ζητούμε συγγνώμη για την ε, καθυστέρηση. Ε, δυστυχώς είχαμε καθυστέρηση ψηφοφορία που έπρεπε να ολοκληρωθεί. Μπας περιπτώσει, τώρα ήρθαμε εδώ και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να έχετε την καλοσύνη ε, πλέον να μην συζητάτε μεταξύ σας και να καθίσετε. Αναφέρουμε και στους συντονιστές. Και όπως ε, πολύ καλά γνωρίζετε, Σήμερα έχουμε μια κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Απασχόλησης και θα συζητήσουμε με τον κύριο Ντομπρόφσκης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος και επίτροπος, αρμόδιος για τον κοινωνικό διάλογο με την κυρία Τάισεν, η κυρία Τάισεν αρμόδια για θέματα απασχόλησης και τον κύριο Μουσκοβισή, ο οποίος είναι αρμόδιος για τα δημοσιονομικά, τη φορολογία, τα τελωνία. Σας καλωσορίζουμε όλου σε αυτήν την κοινή συνεδρίαση. Καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας για τις συστάσεις αναχώρα οι οποίες εγκρίθηκαν από το Σώμα των Επιτρόπων. Ε, υπάρχει μια διαδικασία την οποία όλοι γνωρίζετε ε, θα εγκριθεί από το Συμβούλιο τον Ιούλιο ε, φέτος οι συστάσεις αναχώρα έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί πράγματι αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που καταβάλλεται να υπάρχει μια οριζόντια συνοχή στις ε, συστάσεις αναχώρα έτσι ώστε να λάβουν μια συγκεκριμένη δομή και να δώσουν μια κατεύθυνση στην πολιτική την οποία χαράσει η ευρωπαϊκή πολιτική. Αναφέρομαι στον περίφημο τριγωνικό διάλογο γιατί ε, δεν είναι μόνο ο διάλογος, υπάρχουν πολλά στοιχεία. Οι επενδύσεις, ε, η ε, εξυγίανση, η κοινωνική συνοχή, όλα αυτά τα περιλαμβάνει ο, τριγωνικός, ο τριμερής μάλλον διάλογος και υπάρχει και η αξιολόγηση της ανάγκης να ληφθεί υπόψη γενικότερα το δημοσιονομικό πλαίσιο έτσι ώστε να μπορούμε να εντάξουμε τις ε, προσαρμογές ε, που απορρέουν από τους ε, κανόνες μας. Αυτά με στόχο, όλα αυτά να είναι ευρωϊκά προς την ανάπτυξη, προς την ανάκαμψη, να συμπεριλαμβάνεται επίσης και η κοινωνική διάσταση, η οποία κατέχει ιδιαίτερη σημασία. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στους επιτρόπους για την εισήγησή τους, κύριε Ντομπρόφσκης. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. ότι με πρόεδρε και μέλη του Κοινοβουλίου. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε σήμερα εδώ από κοινού με τους συναδέλφους μου για να σας παρουσιάσω τις συστάσεις αναχώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική πολιτική ε, για τους επόμενους μήνες. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν εξάμεινο αποδείχθηκε ότι είναι το σωστό πλαίσιο για να καθοδηγεί τις προσπάθειες εθνικών μεταρρυθμίσεων η οικονομική μας απόδοση είναι πολύ καλύτερη εφόσον καταβάλλονται οι σωστές προσπάθειες. Η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται και συνεχίζεται σε ανάκαμψη για πέμπτο συναπτό έτος. Ε, είχαμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Ιαπωνία την περασμένη χρονιά. Όλα τα κράτη-μέλη θα αναπτυχθούν, η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανέλθει σε 233 εκατομμύρια πολίτες που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό και αριθμός ανθρώπων που είχε ποτέ απασχόληση και τώρα η πτώχευση βρίσκεται σε καθοδική πορεία η φτώχεια μάλλον. Οι δημόσιες επενδύσεις βελτιώνονται και αυτό το βλέπουμε και σε ε, ε, αριθμό χωρών που βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η, τώρα πλέον ε, για την Πορτογαλία και την Κροατία ολοκληρώθηκε η διαδικασία και έχουμε άλλες οκτώ χώρες, μεταξύ αυτών η Τσεχία, η Δανία και η Σουηδία, οι οποίες χώρες αυτές θα είναι πάνω από τους μεσοπρόθεσμους στόχους και για το 2017 και για το 2018 ως εκ τούτου για τις χώρες αυτές ε, δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη σύσταση αναχώρα για θέματα που να αφορούν σε υπερβολικά ελλείμματα. Δυστυχώς βλέπουμε χώρες οι οποίες αποκλείουν από αυτό το δρόμο προσαρμογής προς το μεσοπρόθεσμο στόχο και γι' αυτό η Ιταλία έπρεπε να λάβει επιπρόσθετα μέτρα 0,2% του ΑΕΠ ε, αυτό το έτος. Επίσης, ε, θέλουμε να δώσουμε συστάσεις στη Ρουμανία για τη σημαντική απόκληση από τον δρόμο της προσαρμογής που ακολούθησε το 2016. Ο Πιέρ θα σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες από αυτού όσον αφορά τα δημοσιονομικά της Ρουμανίας. Βέβαια, η οικονομική ανάκαμψη ε, δεν είναι ισότιμα επιμερισμένη. Ε, ξεκινάμε από την κρίση, είχαμε ε, ανεργία, δημόσιο χρέο σε πολλά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό εξακολουθεί να παραμένει προτεραιότητα. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να χάσουμε το δυναμισμό. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες πρέπει να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές, αντεκτικές. Η ανάπτυξη να περιλαμβάνει όλους τους τομείς, έτσι όλοι να αισθανθούν, όλοι οι πολίτες να αισθανθούν την ανάπτυξη. Και αυτό είναι σημαντικό για να υπάρχει σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτή λοιπόν είναι η στόχη των προσπαθειών μεταρρύθμισης και αυτά συστήνουμε. Οι δικές μας οι συστάσεις ε, ε, διαιρούνται σε τρεις ε, προτεραιότητες ε, και όπως αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο είναι η ανάπτυξη των επενδύσεων, οι διαρθρωτικές αλλαγές και μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Όλα αυτά βεβαίως να προσαρμόζονται σε ειδικέ συνθήκες σε μια συγκεκριμένη χώρα και να έχουν ως στόχο τα θέματα εκείνα τα οποία χρήζουν τις μεγαλύτερες προσοχής αυτό λόγω των μακροοικονομικών δυσκολιών ή και κοινωνικών συνθήκων. Οι χώρες της Ευρωζώνης επίσης εκεί υπάρχουν ειδικέ συστάσεις για την Ευρωζώνη οι οποίε δημοσιεύτηκαν τον προηγούμενο Νοέμβρη. Όσον αφορά τώρα το επίπεδο των συστάσεων, εκεί αντικατοπτρίζεται η κατάσταση και οι προκλήσει που αντιμετωπίζει κάθε χώρα. Και για το λόγο αυτό, χώρε οι οποίε έχουν υπερβολικέ ανισορροπίε, οι χώρε αυτέ θα έχουν πιο λεπτομερεί συστάσει. Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Γαλλία, Ιταλία και Πορτογαλία. Όσον αφορά την Κύπρο, την Ιταλία και την Πορτογαλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αναφέρεται σε συγκεκριμένα προγράμματα εθνικών μεταρρυθμίσεων και συγκεκριμένες διευκρινήσεις έχουν επίσης δοθεί. Υπάρχουν φιλόδοξα σχέδια, ε, δεν υπάρχει λόγος ε, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρχει σωστή και γρήγορη εφαρμογή των ε, μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στις συστάσεις. Εξάλλου έχουμε εντατικοποίησει τον διάλογο με τις κυβερνήσεις, με τα εθνικά κοινοβούλια, με τους κοινωνικούς εταίρους και με άλλους άμεσα εμπλεκόμενους. Καλούμε τα κράτη-μέλη να διαλέγονται με τους ε, εθνικούς ε, συνομιλητές. Εγώ προσωπικά επισκέπτομαι συστηματικά τα κράτη-μέλη και εμπλέκομαι σε συζητήσεις με όλους τους βασικούς φορείς σε εθνικό επίπεδο και το ίδιο πράττουν και άλλοι επίτροποι. Αξιότιμα μέλη. Η ανάπτυξη χωρί αποκλεισμού απαιτεί χρόνο και απαιτεί και ένα μείγμα πολιτική. Χρειαζόμαστε άτομα πολύ καλά εκπαιδευμένα να έχουν και τι απαραίτητε δεξιότητε. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, να αποδίδουμε σημασία επενδύσει επενδύσεις και την καινοτομία. Οφείλουμε να έχουμε κατά νου το εισόδημα και τις ανισότητε οποτεδήποτε σχεδιάζουμε μεταρρυθμίσει. Να στηρίζουμε όσου βρίσκονται σε ανάγκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να καταβάλουν προσπάθειε για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, αλλά η από περιορισμένη πρόοδο μέχρι και ουσιαστική πρόοδο ε, με βάση τις ε, συστάσεις αναχώρα της προηγούμενης χρονιάς. Έχουν ληφθεί πάρα πολλά μέτρα για τη δημοσιονομική πολιτική, για την δημοσιονομική διαχείριση και επίσης και σε σχέση με την πραγματική αγορά. Στο, στην πολιτική προοπτική είχαμε καλύτερη πρόοδο, εκεί περιλαμβάνονται και τα μέτρα τα οποία λήφθησαν λόγω της κρίσης. Υπάρχει λοιπόν πρόοδος, βέβαια η πρόοδος δεν είναι ισομερός καταναμημένη σε όλα ε, σε όλου του τομεί τη πολιτική. Εμεί είμαστε πρότιμοι να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη στην αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τώρα έχουμε ένα σημαντικό εργαλείο, τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, το σχετικό πρόγραμμα στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Βλέπουμε ότι πολλά κράτη-μέλη έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον και έχουν ζητήσει τεχνική βοήθεια. Νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, οι οποίε περιλαμβάνονται και στι συστάσει αναχώρα. Τώρα πλέον η μπάλα βρίσκεται στο κήπεδο των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Μοσκοβισή. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι ε, βουλευτέ κυρίε και κύριοι πρόεδροι. Χαίρομαι που έρχομαι εδώ δίπλα στου συναδέλφου μου και να σα παρουσιάσω με τη σειρά μου ε, το δημοσιονομικό σκέλος του ΕΑΡΝΟΥ πακέτου είναι κάτι που πλέον γνωρίζετε καλά είναι οι προσανατολισμοί τη Κομισιόν για να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη τη Ευρωζώνη να προετοιμάσουν του προπολογισμού του ενώπιση του 2018. Αυτό εγγράφεται στα πλαίσια ενός, μιας οικονομικής και πολιτική συγκυρία συγκεκριμένη σε πολιτικό επίπεδο συνάδει με τη βούλησή μα με τον πολιτικό μα στόχο να δώσουμε μια όθηση στην απασχόληση και την ανάπτυξη και αυτόν τον στόχο έχουμε κατά νου σε αυτή τη φάση ολοκλήρωση του εγγράφου ε, διαβούλευση για το μέλλον τη. Οικονομικής Νομισματική Ένωση. Σε οικονομικό επίπεδο, από ό,τι φαίνεται, συνεχίζεται η οικονομική ανάκαμψη, αλλά αυτή είναι εύθραυστη και κάπω ατυπική, θα έλεγα. Ε, δεν έχουμε φτάσει στι δυνατότητε ε, ανάπτυξη που είχαμε πριν από την κρίση και οι επενδύσει είναι ακόμα χαμηλέ. Το ίδιο ισχύει και για την αύξηση των μισθών. Επίση, παραμένει πολύ χαμηλή η, ε, ο πληθωρισμός παρά την πολιτική, την νομισματική τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει δηλαδή ένα πρόβλημα ζήτηση στην Ευρωζώνη, για να το πούμε σαφώ. Το πακέτο αυτό λοιπόν προτείνει μια έξυπνη εφαρμογή των κανόνων. Είναι σημαντικό η δημοσιονομική πολιτική των κρατών μελών τη Ένωση να βρει το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ τη οικονομική σταθεροποίηση και ε, τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει μέσω επενδύσεων στον τομέα των, ε, των υποδομών ε, θα πρέπει να χρησιμοποιεί, εκεί να πάνε τα χρήματα, όποια περιθώρια υπάρχουν σε δημοσιονομικό επίπεδο. Αυτό το μήνυμα αφορά ε, κυρίως τη Γερμανία και τι κάτω χώρε. Για τα λοιπά κράτη-μέλη θα, πρέπει να χρειαστούν, θα χρειαστούν περαιτέρω προσαρμογές. Να ζητήσουμε όμως ε, πολύ σημαντικέ προσαρμογέ, θα ήταν αντιπαραγωγικό και δεν θα βοηθήσει ούτε την απασχόληση ούτε την ανάπτυξη. Πολλέ αποφάσει έχουν παθεί σε δημοσιονομικό επίπεδο υπό το φω ε, αυτή τη ανάγνωση. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει να κλείσει η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο για την Κροατία και την Πορτογαλία. Εδώ αναγνωρίζουμε τι προσπάθειε που κατέβαλαν ο λαό τη Κροατία και τη Πορτογαλία. δείχνει και την αποτελεσματικότητα των κανόνων μα Είναι ένα καλό νέο, ένα εξαιρετικό νέο για την Ευρώπη. Η, Ευρω... η Ελλάδα τώρα και η Ελλάδα έχει μειώσει ε, το υπερβολικό έλλειμμα κατά το 3% και το 2016 και το 2017. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε και αυτή να βγει από τη διαδικασία υπερβολικού έλλειμματο. Όμω ε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα συζήτηση για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Ε, το Eurogroup, το Eurogroup θα συζητήσει μέσα σε λίγες μέρες και επειδή αυτές οι συζητήσεις για τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας είναι ακόμα ανεξελίξη, η Κομισιόν αποφάσισε να πάρει ε, τη νομική απόφαση και να σταματήσει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος όταν θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση. Αλλά ε, σίγουρα οι παράμετροι για να ακυρωθεί η διαδικασία παραπλοκαλήματος υπάρχουν. Ε, οι συνθήκες πληρώνται. Και αυτό είναι καλό νέο και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Πρέπει να πούμε ότι σε γενικές γραμμές είναι εντυπωσιακή η διαφορά σε σχέση με το 2011. Ε, κάποιοι αμφισβητούν την χρησιμότητα των κανόνων. Υπήρχαν 24 χώρες το 2011 που ήταν σε υπερβολικό έλλειμμα. Ήταν στο 6% το έλλειμμα και σήμερα έχουν μείνει 2-3 χώρες. Ελπίζω το 2018 να μην υπάρχει πια καμία. Και το μέσο επίπεδο ελλείμματος είναι 1,4% το 2017 και προβλέπεται 1,3% για το 2018. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργούν οι κανόνες. Ό,τι αφορά τη Γαλλία και την Ισπανία τώρα. χώρε τη Ευρωζώνης που ακόμα ακολουθούν τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο. Το μήνυμά μα για τι χώρε αυτέ ε, θα επανέλθω και στη συζήτηση φαντάζομαι, είναι ότι η σύσταση του Συμβουλίου στα πλαίσια τη διαδικασία για το υπερβολικό έλλειμμα πρέπει να γίνει σεβαστή. Σε ό,τι αφορά τώρα το προληπτικό σκέλος του συμφώνου, ε, εμείς έχουμε την έκθεση 126.3 όπου εξετάζεται ο μη σεβασμό του κριτηρίου του χρέου για το Βέλγιο και τη Φιλανδία. Για το Βέλγιο η έκθεση φτάνει στο συμπέρασμα ότι σε το στάδιο δεν χρειάζεται να ξεκινήσει μια διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο. Όμω το Βέλγιο θα πρέπει φέτο να πάρει περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα έτσι ώστε να ε, συμμορφώνεται με το σύμφωνο για την περίοδο 2016-2017. Για τη Φιλανδία οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν την αύξηση τη παραγωγικότητα και της απασχόλησης ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν σύντομα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει στη Φιλανδία την απαραίτητη ευελιξία για να μπορέσει να υποστηρίξει αυτή την εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ταυτόχρονα να δοθεί ευελιξία ίδια φύσεω στη Λιθουανία ε, εν ώψη τη εφαρμογή τη μεταρρύθμιση του συνταξιδοτικού συστήματο. Ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση τη Ιταλία, μετά την έκθεση 126.3 που παρουσιάσαμε το Φλεβάρι, η Ιταλία πήρε περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα τη τάξη του 0,2 του ΑΕΠ έτσι ώστε να μπορέσει να συμμορφωθεί με τι υποχρεώσει τη Για την ώρα λοιπόν θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να πάμε παραπέρα στη διαδικασία αυτή. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη δημοσιονομική κατάσταση στην Ιταλία εν ώψη του 2018. Να πω και δύο λόγια για τη Ρουμανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να ζητήσουμε από τη Ρουμανία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα το 2017 έτσι ώστε να διορθώσει τη σημαντική απόκληση που υπάρχει σε ό,τι αφορά την τροχιά προσαρμογής και το δημοσιονομικό στόχο ε, το μεσοποδόσμου του 2016. Είναι η πρώτη φορά που αυτή η διαδικασία τη σημαντική απόκληση εφαρμόζεται. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια προεδοποίηση για να μην ξεκινήσει μια διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο. Και ελπίζουμε οι ρουμανικέ αρχέ ε, να ε, εγκρίνουν αυτά τα μέτρα έτσι ώστε να μην ξεκινήσει η διαδικασία. Το είχαμε πει αυτό και στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ αλλά και στο Eurogroup της περαμένης εβδομάδας. Αυτά κυρίε και κύριοι πολύ πολύ σύντομα το περιεχόμενο στο δημοσιονομικό επίπεδο των συζητήσεών μας. Είμαι δεθειμένος βεβαίως να επανέλθω σε οποιαδήποτε από αυτά τα θέματα στις ερωτήσεις στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μοσκοβισή και τώρα η κυρία Τάισεν έχει το λόγο. Uh, dear President. Πρόεδρε, με του Κοινοβουλίου, η άσκηση φέτος ε, για το εξάμεινο αποτελεί ένα σημείο κατά τεθέν, διότι ε, στην ουσία από την πρώτη ημέρα η προτεραιότητά μας ήταν να αποκαταστήσουμε την ανάπτυξη, την, θέση ε, θέσεις εργασίας και την κοινωνική συνοχή να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα για όλον τον κόσμο. Σήμερα βρίσκομαι εδώ και μπορώ να πω ότι έχουμε διανύσει μεγάλο δρόμο. 233 ε, εκατομμύρια άνθρωποι είχαν απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος. Μεγάλη διαφορά σε σχέση με τρία χρόνια πριν, όπου σε αυτό το διάστημα έχουμε δημιουργήσει πάνω από 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε μια Ευρώπη όπου 90 εκατομμύρια άνθρωποι ψάχνουν δουλειά. Η ανεργία είναι στο 8% που είναι το χαμηλότερο... 19 ε, εκατομμύρια ε, ψάχνουν δουλειά. Η ανεργία είναι στο 8% που είναι το χαμηλότερο επίπεδο. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι έχει μειωθεί η φτώχεια, παρόλα αυτά παραμένει ψηλά. Η ανισότητες αποτελούν μεγάλο ε, πρόβλημα και ανησυχία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι επηρεάζουν τον κοινωνικό ιστό, τις οικονομικές προοπτικές και γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν έχει επικεντρωθεί ακριβώς σε αυτό το ζήτημα της κοινωνικής συνοχής. Πρώτον, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ξεκάθαρο στην ανακοίνωση που ε, συνοδεύει τις στάσεις για την αναχώρα για το 2017 ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη τον κοινωνικό αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων τους ε, στην, ε, στο σχεδιασμό, στην αλληλουχία των μεταρρυθμίσεων και στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Ζητούμε λοιπόν από τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι οι μεταρρυθμίσεις ε, προωθούν την κινητικότητα και μειώνουν τις ανισότητες αντί να τις επιδεινώνουν. Επίσης η Κομισιόν ε, θέτει ε, στο επίκεντρο ε, τον κοινωνικό πυλώνα, ο οποίος ε, δίνει έμφαση στην πάταξη των ανισοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, λοιπόν, έχει γίνει σημαντικό εργαλείο για να μπορέσει αυτός ο πυλώνας να τεθεί σε εφαρμογή. Υπάρχουν, λοιπόν, οι συστάσεις ε, που μας δίνουν ακριβώς την κατεύθυνση. Παράδειγμα, η πρώτη αρχή είναι η σημασία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της διαβίου μάθησης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι στην Ευρώπη θα έχουν πρόσβαση στις καλύτερες ευκαιρίες μάθησης. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα οριστεί και θα οριστούν και οι πιθανότητε που έχουν να επιτύχουν στη ζωή του. Η ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη, διότι οι επιχειρήσει μα χρειάζονται ταλέντο για να ευημερήσουν. Θα πρέπει λοιπόν να, να βοηθήσουμε του ανθρώπου, να αποκτήσουν περισσότερε δεξιότητε ή να αλλάξουν την κατεύθυνση των δεξιοτήτων τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Επίσης θέλουμε να δώσουμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια. Αυτό παραμένει προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ο να τονίζει τη σημασία των ε, δίκαιων μισθών που θα διασφαλίσουν ένα καλό βιωτικό επίπεδο. Αυτό είναι στις συστάσεις ε, που αναφέρονται στην οικονομική ανάπτυξη και στα δικαιώματα των εργαζομένων για κάποιες χώρες. Ε, όλα αυτά βέβαια με την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον κοινωνικό διάλογο όποτε χρειάζεται. Φυσικά ο πυλώνας ζητά συστήματα κοινωνικής προστασίας που θα αποτελούν μια ε, επένδυση στους ανθρώπους της Ευρώπης. Θέλουμε με τη συστάση μας να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες με πιο επαρκή συστήματα κοινωνικής προστασίας και καλύτερη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη, μακροχρόνια περίθαλψη και φροντίδα των παιδιών. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ, διότι με τις σκληρές μας προσπάθειες καταφέραμε να έχουμε θετική στροφή από το 2013 και μετά. Μπορεί να υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να έχουμε μια ανάπτυξη που θα τους περιλαμβάνει όλους στην Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην ουσία αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς για να το πετύχουμε αυτό και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι το κλειδί που θα μας οδηγήσει ε, σε αυτή τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο. Οι εθνικές ε, κυβερνήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι, οι κοινωνικοί κοινωνία γενικά θα πρέπει τώρα να πάρει τη σκητάλη και να μας βοηθήσει να έχουμε μια πιο ευημερούσα κοινωνική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε τώρα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Για να αντιμετωπίσουμε την καθυστέρηση προτείνω να τις συγχωνεύσουμε σε μπλοκ ερωτήσεων. Θα κάνουμε δύο μπλοκ ερωτήσεων. Να υπογραμμίσω απλώς αυτό που είπε ο Πιέρ Μοσκοβής στην ΣΥ για την αποτελεσματικότητα των κανόνων όταν αυτοί εφαρμόζονται και με έξυπνο τρόπο, το προσυπογράφω. Βλέπουμε εδώ τρεις χώρες από τις 24 στο 0 ίσως 1,3% του ελλείμματος. Πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα Γκούναρ είναι ο Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που ακούσαμε. Ε, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να καλωσορίσουμε βέβαια το γεγονός ότι τα πάμε καλύτερα, αλλά το ότι τα πάμε καλύτερα δεν σημαίνει ότι τα πάμε όσο καλά θα έπρεπε. Ε, βιώνουμε μια ανάκαμψη και αυτή είναι σε γενικότερο επίπεδο, συνολικά. Δηλαδή, Ξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Αν έχει κανείς το κεφάλι στο φούρνο και το, τα πόδια ή αντίστροφα στο ψυγείο, υπάρχει μια μέση καλή ε, θερμοκρασία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η ε, κατάλληλη. Θέλω λοιπόν να πω ότι καταρχήν η ανάπτυξη κατά κεφαλή είναι πάρα πολύ μικρή. Και το δεύτερο, σε ορισμένα κρατημέλη δεν υπάρχει ικανοποιητική ανάπτυξη. Απόλυτα μη ικανοποιητική. Το 8% ανεργία σημαίνει ότι έχουμε υψηλότερη ανεργία σε αρκετά κρατημέλη από ό,τι θα έπρεπε και ορισμένοι άνθρωποι ούτε καν καταγράφονται, είναι εκτός αγοράς εργασίας. Άρα δηλαδή πρέπει να υπάρξουν υψηλότερα μέτρα, να ανέβει ο πύχης για την ανάπτυξη. Περί αυτού πρόκειται. Και θα ήθελα καταρχήν να απευθυνθώ στον Επίτροπο κ. Ντομπρόφσκη, αλλά και στους ε, κυρίους ε, Μοσκοβισή και στην κυρία Τάισεν και να ερωτήσω το εξή. Πώ μπορούμε να θέσουμε υψηλότερου στόχου καταρχήν για δυνάμια ανάπτυξη. Η κοινωνική συνοχή σημαίνει καταρχήν διαρθρωτική συνοχή και αυτό που διαπιστώνουμε στι διαφορέ που υπάρχουν στι οικονομίε μα είναι ότι εφαρμόζονται διαφορετικά επίπεδα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Νομίζω λοιπόν ότι και εσεί θα πρέπει να είστε περισσότερο ευθύ επ' αυτού. Όχι μόνο να μιλάτε έτσι γενικά ότι χρειάζονται διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, αλλά να γίνουν μεταρρυθμίσει στι χώρε εκείνες όπου υπάρχει χαμηλότερη πραγματική και ενδυνάμια ανάπτυξη. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο να γίνουν περισσότερα. Και θα ήθελα παρακαλώ να μας ενημερώσετε, να τοποθετηθείτε επ' αυτού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι όντως μια σημαντική στιγμή, η στιγμή των συστάσεων αναχώρα, διότι θεωρητικά θα επιτρέψει να συμφιλειώσουμε δύο στόχους. Η ανάκαμψη με επενδύσεις και ανάπτυξη ε, και τα δημοσιονομικά. Αφενός λοιπόν έχουμε τους σχέδιο επενδύσεων που φέρνει κάποια αποτελέσματα, αλλά οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμένουν χαμηλοί. Παραμένουν χαμηλοί για να μειώσουμε την ανεργία την οποία γνωρίζουμε ή για να τη μειώσουμε τουλάχιστον σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Οι δύο αυτοί στόχοι, δηλαδή οι επενδύσεις, η ανάπτυξη αλλά και ο έλεγχος δημοσιονομικών, ε, έχουν επιπτώσεις αντιφατικές. Εάν δούμε τις συστάσεις που γίνονται για τη χώρα μου, το Βέλγιο παραδείγματος χάρη, η Κομισιόν σωστά λέει ότι είναι χαμηλή η ποιότητα των υποδομών. Αλλά αυτή η χαμηλή ποιότητα των υποδομών είναι αποτέλεσμα υποεπένδυσης που σχετίζεται με τα μέτρα ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης. Αυτή την αντίφαση την ξαναβρίσκουμε και στο επίπεδο της κατάρτισης, της εκπαίδευσης, ε, στον τομέα ε, των επενδύσεων στην έρευνα, αλλά και στις κοινωνικές πολιτικές. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς μπορούμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την αντίφαση μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων. Υπογραμμίζω βεβαίως την ικανοποίησή σας να... την ικανοποίηση την βούλησή σας να γίνει μια προσπάθεια να μειωθούν οι ανισότητες. Το έχω ξανακούσει, αλλά θα ήθελα να μου πείτε πώς θα ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος. Ο κοινωνικός διάλογος είναι απαραίτητος για την κοινωνική συνοχή. Τι θα κάνετε για να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό έχει ο καθένας. Η κυρία Περφόνς Μπέρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία την Πρόεδρε, κυρία Επιτροπή. Σας ευχαριστώ ε, για αυτήν την ε, έτσι κάπως γαλήνια απεικόνηση της κατάστασης ε, σε ό,τι αφορά τις συστάσεις αναχώρα στα εργαλεία που έχουν να κάνουν με που έχουν τα κράτη-μέλη στη διάθεσή του, υπάρχει ένα μεταξύ των εργαλείων αυτών που έχει να κάνει με τον καλύτερο συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το εργαλείο τη φορολογία. Πολλέ από τι μεταρρυθμίσει που ζητάτε από τα κράτη-μέλη περνούν από την εξέλιξη των φορολογικών πολιτικών στα κράτη-μέλη και βλέπω ότι για κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν κάποιε συστάσει ε, ή θα μπορούσαν να γίνουν κάποιε συστάσει για τα φορολογικά. Ε, θα ήθελα να ξέρω πώς βλέπετε εσείς τα κράτη-μέλη ε, να κάνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις ε, οι οποίες θα οδηγούν σε μια μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ φορολόγησης του κεφαλαίου και της εργασίας διότι υπάρχουν πολλές συστάσεις που ανησυχούν για το ύψος της φορολόγησης στις χαμηλές, ε, στους χαμηλούς μισθούς. Ε, ταυτόχρονα έχουμε τη φορολόγηση που ε, είναι υπέρ του χρέους και τη φορολόγηση που δεν πάει προς την κατεύθυνση αυτή. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό το θέμα της φορολόγησης και θα πρέπει να έχει αντίκτυπο στις πολιτικές μας. Η Μαρία Αρένα έχει τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον Ζόρζο Ρολάν για τα αντιφατικά στοιχεία που αναφέρθηκαν πριν, γιατί θα μπορούσαμε να βγούμε από την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος σε κάποιες περιπτώσεις, όμως το ερώτημα είναι ποια είναι η σχέση μεταξύ των μέτρων αυτών που είναι δημοσιονομικά μέτρα και της επιδίνωσης ε, της κατάστασης της κοινωνικής στην Ευρώπη σήμερα. Έχουμε επαρκείς δείκτες για να μας δείξουν αν μια χώρα που βγαίνει από το υπερβολικό έλλειμμα μπορεί να αντιμετωπίσει σωστά και την κατάσταση των ανισοτήτων. Κατανοώ την ε, θέληση του συναδέλφου να πάμε περισσότερο προς την πάταξη της φτώχειας στην Ευρώπη, όμως ε, η επαγγελματική ζωή, ε, η ευελιξία των θέσεων εργασίας ε, μας οδηγούν στη σωστή κατεύθυνση, γιατί θεωρώ ότι οδηγούν στη φτώχεια και κυρίως ε, στη γυναικεία ε, φτώχεια. Είναι ένα θέμα λοιπόν που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα που έχουν οι γυναίκες σε επίπεδο φτώχειας, ειδικά στις πιο φτωχές χώρες. Όταν μιλάμε για επενδύσεις, ε, ε, μιλάμε, δεν μιλάμε για αυτές που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή μετάβαση, οι οποίες θα φέρουν πολλές, που θα φέρει πολλές θέσεις εργασίας ε, και βοηθούν γενικότερα στην οικοτομία. Ευχαριστώ. Παίρνει το Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μια ερώτηση προς τον κύριο Ντομπρόφσκης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πολλωστή φορά επικρίνει το υπερβολικό πλεόνασμα της Γερμανίας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, ε, σε ποια οικονομική ανάλυση βασίζεστε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ε, ξέρω, σας ε, απασχολεί το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ή σας απασχολεί το πλεόνασμα στο εμπόριο με προϊόντα και με υπηρεσίες. Αναφέρεται ότι η Γερμανία θα πρέπει να αυξήσει τις δημόσιες επενδύσεις και θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι στη Γερμανία οι δημόσιες επενδύσεις θα οδηγούσαν στο ότι οι γερμανικές εταιρείε θα περιόριζαν τις εξαγωγές, θα είχαν λιγότερες εξαγωγές σε άλλες χώρες. Ή μήπω πιστεύει η Επιτροπή ότι οι εισαγωγέ προς τη Γερμανία θα αυξάνονται σημαντικά αν εφαρμόζονταν επενδυτικά προγράμματα στη Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πρόκειται τόσο για το πλεόνασμα στο ιδιωτικό εμπόριο με ε, προϊόντα και ε, συναλλαγές, αλλά την ενδιαφέρει περισσότερο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η Γερμανία λοιπόν όπως γνωρίζετε, έχει επιτύχει και έσοδα από δανειοδότηση σε τρίτες χώρες και ερωτώ, τι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε εάν οι εσωτερικές καταθέσεις χρησιμοποιηθούν περισσότερο ως επενδύσεις και όχι ως δάνεια σε τρίτες χώρες. Η Ουλούρη Τρεμπέτσιους, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς ο ίδιος ε, είπατε ότι κατ' ουσίαν κάθε κράτος μέλος ε, χρειάζεται μια δική του πολιτική πρωτοβουλία έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα διέξοδα. Εσείς ο κύριος Ντομπρόφσκης μιλήσατε για συστάσεις ε, κομμένες και ραμμένες ε, στις ανάγκες μιας χώρας. Βεβαίως αυτό που κατέστη απόλυτα σαφές είναι ότι δεν υπάρχει μια τέτοια μαϊκή συνταγή one size fits all διότι κάθε κράτος μέλος αντιμετωπίζει και διαφορετικές προκλήσεις και αναφέρεστε στον κοινωνικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν τα κανείς αυτά θα έχει την υποψία ότι καταβάλλεται η προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταφέρει ένα κοινωνικό διάλειμμα, θα το χαρακτήριζα, σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση λένε πολύ, έχει πολύ ψηλέ κοινωνικέ προδιαγραφές, καλό αυτό, αλλά θα πρέπει κανείς και να μπορεί να τις χρηματοδοτεί. Ε, τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να βρουν και κάποιες δυνατότητε να εφαρμόζουν στην πράξη συγκεκριμένα μέτρα. Όσο έχει λοιπόν η οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υπερβολικές κοινωνικές απαιτήσει είναι κίνδυνος. Βεβαίως, ε, κάποια πλούσια κρατημέλη έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν υψηλότερες κοινωνικές προδιαγραφές, έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν κανόνες, όμως υπάρχουν και πιο αδύναμες χώρες. Εσείς ο ίδιος τις ονοματίσατε Παραδείγματο χάρη στην Ανατολική Ευρώπη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίε είναι η σπονδυλική στήλη τη οικονομία μας, Αυτέ οι επιχειρήσει δεν μπορούν να εφαρμόσουν αυτέ τι υψηλέ κοινωνικέ προδιαγραφέ. Και σα ερωτώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προτίθεται να εφαρμόζει αυτόν τον κοινωνικό πυλώνα και παράλληλα να διατηρείται η υπευθυνότητα των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, και ο Καλβέ Σόμπο. Κάθε εξάμεινο έχουμε την τιμή να συναντούμε τους τρεις αυτούς εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Χαιρόμαστε βέβαια που βλέπουμε από οικονομικής πλευράς πολλές χώρες ε, έχουν ε, μπει στο δρόμο αυτό δεν ισχύει για τη χώρα μου, ούτε για την εκλογή μου περιφέρεια, αλλά εν πάση περιπτώσει θα επανέλθουμε. Πολύ αργά βέβαια προχωρούν όλα αυτά, πολύ ε, ε, 2% αριθμοί ανάπτυξη δεν είναι εκεί για να πανηγυρίζουμε, ιδιαίτερα όταν αυτή η ανάπτυξη είναι κατανεμμένη πολύ άνισα και βεβαίω υπάρχουν σημαντικά διαθροτικά προβλήματα. Ε, άκουσα για παραγωγικότητε, άκουσα παραγωγικότητα και για ανισότητε. Ε, και ότι πρέπει να πάρουν πιο σημαντική θέση. Ιδιαίτερα το θέμα των ανισοτήτων που αυτή τη στιγμή καταστρέφουν την πολιτική μας, το πολιτικό μας κεφάλαιο, την πολιτική υποστήριξη που μπορεί να έχουμε. Χαίρομαι που άκουσα λοιπόν για ανισότητες, αλλά θέλω να δω και κάτι πρακτικό. Επίσης η Κομισιόν ε, θα πρέπει να πάει λίγο πιο μακριά σε διαθροτικό επίπεδο. Είναι πολύ βραχή η με προσέγγιση της. Είναι βασισμένη ε, σε ποσοτικά στοιχεία ε, μόνο. Βεβαίως ε, τα κράτη-μέλη ουσιαστικά προσπαθούν να ξεγελάσουν την Κομισιόν και κοσμένες φορές ε, η Κομισιόν ορισμένες φορές πέφτει στην παγίδα. Παραδείγματος χάρη ζητάει από τη δική μου εκλογική περιφέρεια να έχει έναν σταθερό προπολογισμό. Πολύ ωραία. Όταν λοιπόν παρουσιάσουμε ένα προπολογισμό με στοιχεία ισορροπημένα είναι ευχαριστημένη η Κομισιόν. Με αυτό το προπολογισμό όμως έχουν προκύψει πολύ σημαντικέ ανισότητε στην Ισπανία που θα δημιουργήσουν ε, στο μέλλον δημοσιονομικά ελλείμματα ε, στη χώρα μου. Θα πρέπει λοιπόν να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις διαθροτικές πτυχές και να μην την ξεγελούν οι αριθμοί. Και επίσης θα ήταν καλό να το δείτε πιο μακροπρόθεσμα το θέμα, πέρα από το εξάμεινο. Αν έλαβα χώρα όντως διαθροτικές μεταρρυθμίσεις, ε, αν όντως φτάνουμε στην παραγωγικότητα. Υπάρχουν χώρες όπου η ενεργειακή πολιτική ε, την οδηγεί ε, στο να είναι φτωχή και να έχει ενεργεία για δεκαετίες. Ε, ήθελα να πω επίσης ότι η μόνη λιτότητα που κάνει κακό στην Ευρώπη είναι η γερμανική. Διότι οι Γερμανοί πρέπει να επιτρέψουν στους πολίτες να ζήσουν καλύτερα, να ξοδέψουν περισσότερα και καλύτερα. Μπορούν και έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Αν πω, Πήρατε και το χρόνο άλλων συναδέλφων που δεν είναι εδώ, οπότε μπορούμε τώρα να έχουμε τις πρώτες απαντήσεις από τους επιτρόπους. Ποιος θέλει να ξεκινήσει, ο κύριος Δομπρόφσκης. Ευχαριστώ συνάδελφοι για τις ερωτήσεις. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια από τα θέματα που τέθηκαν αναομάδες. Καταρχάς, όντως, στο θέμα που θέσατε για τα συνολικά νούμερα και για τις ε, διαφορές και ανισότητες που μπορεί να κρύβουν, ε, όντως υπάρχουν διαφορές σε επίπεδο ποσοστών ανάπτυξης ε, αλλά και ανεργίας. Εμείς θέλουμε όμως και βλέπουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα έχουν ανάπτυξη φέτος. Βέβαια δεν είναι ίδια τα επίπεδα της ανάπτυξης σε κάθε χώρα σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων που αντιμετωπίζουν τα διαρθρωτικά προβλήματα των κρατών μελών, όπως ας πούμε ε, τα χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης. Ε, είδα, είπα ήδη ε, ότι υπάρχει η διαδικασία μακροοικονομικής αστάθειας, υπάρχουν εξαιρετικές αστάθειες, ανισότητες, οι οποίες συνήθως αποτελούν αντικείμενο πιο συγκεκριμένων συστάσεων και ενός μηχανισμού παρακολούθησης για κάποιες χώρες. Είναι οι αρχές που αναφέρατε και εσείς, ότι χρειάζεται να εργαστούμε περισσότερο προς την κατεύθυνση της επίληψης ε, των μεγαλύτερων διαρθρωτικών ε, προβλημάτων. Στη συνέχεια, για το πώς ε, θα δούμε, ε, πώς θα συνδυάσουμε τις ανάγκες ε, για περισσότερες επενδύσεις με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, αλλά και την δημοσιονομική προσαρμογή που πρέπει να επιδιώξουν πολλά κράτη-μέλη. Το έθεσαν πολλοί ευρωβουλευτές. Όντως, πρόκειται για ένα ζήτημα που πρέπει να γνωρίζουμε και ένα θέμα που πρέπει να θέσουμε σε ισορροπία. Και το έχουμε τονίσει φέτος το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και στις ε, συστάσεις αναχώρα. Ειδικά στο δημοσιονομικό επίπεδο. Φυσικά, αξίζει να σημειώσουμε ταυτόχρονα ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας απλώς και μόνο συσσωρεύοντας περισσότερο χρέος Υπάρχουν υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους σε πολλέ ε, χώρες και αυτό είναι μια διαρθρωτική αδυναμία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει λοιπόν τα δημοσιονομικά να είναι βιώσιμα και να έχουμε και ξεκάθαρη μείωση των προβληματικών στοιχείων σε σταθερή βάση. Τώρα για τον κοινωνικό πυλώνα και τα μέτρα στην αγορά εργασίας ε, θα απαντήσει η Μαριάν τα ζητήματα που τέθηκαν σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι και πάλι ένα θέμα το οποίο τονίστηκε φέτος στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ε, μιλάμε για την ε, συνολική δημοσιονομική κατάσταση ε, στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη συγκεκριμένα και στα κράτη της Ευρωζώνης συστάσει αναχώρα για τη φορολογία τώρα. Η γενική μας ε, συμβουλή είναι να μειώσουμε την φορολογία της εργασίας, ειδικά των χαμηλομίσθων, διότι αυτή η προσέγγιση είναι η επιθυμητή και την παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Επίσης, ε, στα πλαίσια της πρότασης της CTB έχουμε ε, ζητήματα που αφορούν ε, στις, ε, στα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων, τα οποία καλύπτουν την ίδια πτυχή. Τώρα, το παραδοσιακό ερώτημα για το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαχών της Γερμανίας. Αυτός είναι και ο λόγος που η Γερμανία είναι ε, στη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, διότι υπάρχει αυτό το πλεόνασμα. Είναι 6% του GDP παραπάνω από το σημείο αναφοράς. Είναι μία τάση η οποία έχει διατηρηθεί για πολύ χρονικό διάστημα. Συνεπώς, ε, συστήνουμε να ενισχυθεί η πλευρά της ζήτησης στην οικονομία, να ενισχυθούν οι επενδύσεις Μιλήσατε και για τις εισαγωγές-εξαγωγές μεταξύ άλλων. Μέσα από την ενίσχυση της ζήτησης ε, και της επενδύσης ε, περιμένουμε ότι θα έχουμε και υψηλότερη αύξηση των ε, εισαγωγών. Δεν σημαίνει βέβαια ότι εμείς θέλουμε να έχουν λιγότερες εξαγωγές οι γερμανικές επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό που συστήνουμε. Όπως και να έχει όμως, ε, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η Γερμανία ήδη έχει κάνει περαιτέρω επενδύσεις. Ήδη από πέρυσι υπήρξε πρόοδος σε αυτόν τον τομέα. Παραμένει όμως το πλεόνασμα τρέχουσών συναλλαγών, του συζυγίου τρέχουσών συναλλαγών πάνω από το επίπεδο αναφοράς. Τέθηκε επίσης ε, το θέμα ε, του ότι δεν υπάρχει μία λύση μαγική για όλους. Ε. Και πάλι αυτή η ερώτηση έχει να κάνει με τον κοινωνικό πυλώνα και η Μαριάννα θα την απαντήσει. Όμως εμείς είμαστε ξεκάθαροι δεν θέλουμε νέες αρμοδιότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κοινωνικό τομέα. Αυτό θα παραμείνει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, κατά κύριο λόγο. Ένα ερώτημα επίσης τέθηκε σχετικά με την ανάπτυξη της παραγωγικότητας, ε, την μείωση των ανισοτήτων, τα πρακτικά μέτρα που επιζητούμε. Τα μέτρα λοιπόν που προτείνουμε στα κράτη-μέλη, στις συστάσεις αναχώρα φυσικά, διότι αν δείτε γενικά, ε, τις συστάσεις αναχώρα, αυτό ακριβώς δίνουμε πρακτικά μέτρα που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας, στην αγορά των υπηρεσιών, στην ε, βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και ούτω καθεξής. Ως προς την ανισότητα, μιλάμε για την φορολογική πολιτική, για καλύτερη στόχευση στα κοινωνικά συστήματα, οι δεξιότητες, ε, ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, όλα αυτά τα στοιχεία θα μειώσουν την ανισότητα. Σε Ευχαριστούμε κύριος Μασκοβησί. Πολύ σύντομα, ε, συμφωνώ με τα πρώτα πρα, την πρώτη παρέμβαση του κυρίου Μάρκ ότι βεβαίως πάνε καλύτερα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι πάνε και καλά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να επαναπαυόμαστε. Είναι ακόμα ισχνή η ανάπτυξη σε σχέση με την παγκόσμια ανάπτυξη τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλά, οι ανισότητες επίσης είναι εντυπωσιακέ. Το ζήτημα είναι λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την, τους ρυθμούς ανάπτυξης. Και υπάρχουν εδώ τρία θέματα που τίθενται. Αφενός πρέπει να συνεχίσουν, να συνεχιστούν οι διαστατικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό ισχύει για όλους. Ιδιαίτερα ε, οι χώρες βέβαια που είναι κάπως πιο πίσω να μειωθούν οι μακροοικονομικές ανισότητες και εδώ συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις στις χώρες όπου, αυτό είναι εφικτό και τρίτον να μειώσουμε τις αποκλίσεις στην Ευρωζώνη. Συνδέεται αυτό και με το πρώτο ζήτημα. Είναι και ένα από τα θέματα της Λευκής Βίβλου που θα υποβάλουμε για την ε, εμβάθυνση της Ευρωζώνης. Εάν έχουμε όλο και μεγαλύτερες αποκλίσεις στην Ευρωζώνη, ακόμα και με την προστασία του ευρώ, ε, κάποια στιγμή θα τεθεί ένα θέμα ε, δημοκρατικής νομιμότητας, ε, πολιτικό θέμα. Γι' αυτό λοιπόν η εμβάθυνση της Ευρωζώνης θα πρέπει να οργανωθεί γύρω από αυτήν την έννοια της σύγκλησης, της μακροοικονομικής σύγκλησης. Και τα μέτρα που θα πάρουμε, όλα τα μέτρα, είτε αφορούν τη δημιουργία ε, μιας δημοσιονομικής ε, δυνατότητας ε, ή είτε αλλάξει ο τρόπος ε, διακυβέρνησης. Πρέπει να έχουν κατά νου αυτό τον στόχο. Τώρα, μιλάμε αφενός, μιλάμε για μια αντίφαση μεταξύ επενδύσεων και δημοσιονομικής εξυγίανσης. Προσοχή, υπάρχει το θέμα της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών. Εγώ δεν νομίζω ότι το να εξηγιάνουμε, να μειώσουμε τις ελλείψεις, ε, τα ελλείμματα, ε, αυτό είναι εις βάρος των επενδύσεων. Είναι θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων, πολιτικού προσανατολισμού. Πιστεύω ότι σαφώς θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις για όλες τις χώρες. Για τις χώρες που έχουν δυνατότητες λόγω πλεονασμάτων, αλλά και για τις άλλες. Βεβαίως σε κάποιες χώρες ε, εμφανίζονται εμπόδια στις, στις επενδύσεις αυτές, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όμως η Κομισιόν σίγουρα είναι υπέρ των επενδύσεων. Ήταν και το νόημα του σχέδιου Juncker που έχει στεφθεί από επιτυχία. Ε, έχουν ε, διατεθεί πάνω από 100 δισεκατομμύρια ε, ευρώ έως τώρα. Η κυρία Μπερέζ είπε πολύ σωστά ότι αναφέρθηκε στο θέμα της φορολόγησης των μικρών εισοδημάτων, των χαμηλών εισοδημάτων. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε για τα φορολογικά εργαλεία που είναι υπέρ του χρέους Υπάρχουν δύο σχέδια της Κομισιόν. Καταρχήν ε, η Ένωση των Κεφαλαίων και μία ενιαία φορολογητέα βάση για τον, για τον φόρο επιχειρήσεων. Είναι ένα σχέδιο πολύ σημαντικό, δομικό, το οποίο προσπαθούμε να προωθήσουμε και, είναι, και έχει πολλές λειτουργίες καταρχήν απλοποιεί ε, πολύ σημαντικά σε φορολογικό διοικητικό επίπεδο, μειώνει την επιβάρηση των επιχειρήσεων, ταυτόχρονα είναι ένα καταπληκτικό ε, εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της φορολογικής απάτης και της φορο, ε, φοροδιαφυγής και ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη με από την αποτυχία του παρελθόντος, ε, θέλουμε να δώσουμε κάποια κίνητρα ε, για τις επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης, της καινοτομίας και ό,τι συνεισφέρει στην ε, ανάπτυξη της ισοτιμίας. Ε, είναι κάτι λοιπόν που ζητούμε από το Συμβούλιο. Η πρώτη συζήτηση λοιπόν ε, στο ΕΚΟΦΗΝ είχε αυτή την, το αντικείμενο με σημαντική υποστήριξη από τα κράτη-μέλη αλλά και με δισταγμούς από κάποια άλλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοιχτή βεβαίω σε συμβιβασμού. Αλλά πρέπει να είναι συμβιβασμοί ποιοτικοί. Αλλιώ δεν είναι συμβιβασμοί, είναι ε, εγκατάλειψη μια προσπάθεια. Θα πρέπει λοιπόν να φτάσουμε μέχρι το τέλο τη προσπάθεια αυτή. Και για να απαντήσω και στην κυρία Αρένα, μπαίνουν τα ζητήματα της ποιότητας των τη δημόσια χρηματοδότηση. Διότι δίνουμε όντω μεγάλη έμφαση στα ποσοτικά στοιχεία, στον έλεγχο των ελλείμματων βεβαίω, αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να ελέγξει κάποιο τα ελλείμματα και ο καλύτερο τρόπο είναι να δοθεί έμφαση στην ποιότητα των δημοσίων επενδύσεων, των δημοσίων δαπανών και αυτό πρέπει ταυτόχρονα βέβαια να συνεισφέρει και στην μείωση των ανισοτήτων. Ευχαριστώ. Η κυρία Τάισεν. Uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά στην ερώτηση του κύριου Χόκμαρκ, ε, δηλαδή το πώς μπορούμε να οργανώσουμε τα συστήματά μας ε, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη γιατί αυτή που υπάρχει τώρα δεν αρκεί. Όσον αφορά τα δικά μου τα θέματα εμείς υπό τον κοινωνικό πυλώνα και υπό το θεματολόγιο των δεξιοτήτων, ισχυριζόμαστε ότι θα πρέπει να οργανώσουμε την αγορά εργασίας με ίδιο τρόπο, έτσι ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτή την αγορά και να μπορούν να αναπτυχθούν οι δεξιότητες και τα προσόντα. Όλοι να έχουν πρόσβαση στην καλή παιδεία. Η παιδεία είναι πολύ σημαντική, να μπορούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν περαιτέρω οι δεξιότητες. Οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα Διαβιωμάτιση όχι μόνο όταν θα είναι 25 αλλά και όταν θα είναι 55 και 60 ετών γιατί θέλουμε να παραμείνουν περισσότερο στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να τονώσουμε τις δεξιότητες για να έχουμε καλύτερη παραγωγικότητα και δυνατόν και καινοτομία. Ο κύριος Κλώτρολό έκανε θετικές, ε, θετικά σχόλια για τον αγώνα μας κατά της ε, ανισότητας και τέθησαν και ερωτήματα σχετικά με τον κοινωνικό διάλογο. Τι δηλαδή κάνουμε για να βελτιωθεί και να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος. Γνωρίζετε ότι η Επιτροπή ανέλαβε τότε είχαμε αυτό που αποκαλούμε συνδιάσκεψη ψηλού επίπεδου, διότι εκεί συμμετείχαν πολλοί από τους κοινωνικούς εταίρους και όλοι συμφωνήσαμε ότι θα ενισχύσουμε τον κοινωνικό διάλογο και αναλάβαμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Η μία ήταν να υπάρχουν περισσότερες διαβουλεύσεις ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όχι μόνο αυστηρά για κοινωνικές αλλά και για άλλες πολιτικές που είναι καθοριστικές για την οικονομία και γενικότερα για την κατάσταση της κοινωνίας. Και αυτό πράττουμε. Τώρα λοιπόν διεξάγουν περισσότερες διαβουλεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα στα, στους κοινωνικούς εταίρους, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σας είπα, αλλά και σε επίπεδο εθνικό. Εξάλλου, αυτό επί το οποίο συμφωνήσαμε και δουλεύουμε πάνω σε αυτό είναι να ε, προωθήσουμε τις δεξιότητες επίπεδο κρατών μελών. Αυτό ε, είναι εν το γίγνεσθε, είναι μια δουλειά χρονοβόρα, ε, δεν μπορεί να πει κανείς, α, αποφάσισα πάτη στα κουμπί και να οι δεξιότητε. δεν πάει έτσι. Ε, όλα έχουν σχέση με την ε, αντιπροσωπευτικότητα, παραδείγματο χάρη. Εμείς ως ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήξαμε στο ότι χρειαζόμαστε τους κοινωνικούς εταίρους για το σχεδιασμό των πολιτικών μας. Αν οικειοποιηθούν οι εταίροι τα προγράμματα, θα καταλαβαίνετε ότι μπορούν να προχωρήσουν και πολύ καλύτερα. Όσον αφορά τώρα στο θέμα της φτώχειας της Μαρία Ρένα, ε, η φτώχεια και η κατάσταση των γυναικών στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να πω ότι όταν μιλάμε για την ευελιξία, για τη μερική απασχόληση, είναι αλήθεια ότι πολλοί ε, θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερο. Όμως, πολλοί εξ αυτών, μην ξεχνάτε, είναι και ευτυχείς. Ως εκ τούτου, η ευελιξία στις ρυθμίσεις εργασίας έχει αποδείξει ότι μπορούμε να βοηθήσουμε ε, γονείς, γυναίκες, Εντάξει, δεν λέω πάντα, μερικέ φορέ. Είμαι πολύ προσεκτική στη διατύπωσή μου, γιατί γνωρίζουμε ε, και γι' αυτό σας παρουσιάσαμε και πριν από μερικές εβδομάδε αυτό το πακέτο της διαβίου μάθησης, Γνωρίζουμε ότι πολλές γυναίκες που έχουν παιδιά και άλλους για τους οποίους ε, μεριμνούν. Η συμμετοχή των γυναικών αυτών στην αγορά είναι περιορισμένη, εργάζονται με μερική απασχόληση γιατί μπορούν να συνδυάσουν πολλά πράγματα. Βέβαια, τα εισοδήματά τους είναι πολύ χαμηλότερα και αυτό επηρεάζει όχι μόνο το επίπεδό τους, αλλά και την μελλοντική τους συνταξιοδότηση. Και γνωρίζουμε όλο ε, πόσο σημαντικό είναι το χάσμα στους μισθούς και στις συντάξεις. Γι' αυτό λοιπόν να υπάρχει ισορροπία και όπως σας είπα στο πακέτο της διαβίωματσης. υπάρχουν και άλλες διατάξεις μη νομοθετικές. Στο πλαίσιο του εξαμήνου έχουμε τονίσει ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχουν καλύτερες εγκαταστάσεις μέρημνας για τα παιδιά έτσι ώστε να μπορούν όλοι να συνδυάσουν καλύτερα την ιδιωτική του ζωή με την εργασία τους. Ε, για τη φτώχεια γενικά γνωρίζετε κι εσείς ότι πρόκειται για ένα πολυδιάστατο πρόβλημα. Δεν είναι ότι με ένα μόνο πράγμα μπορεί κανείς να λύσει το πρόβλημα. Πρέπει να δουλέψουμε και στα τρία επίπεδα του πυλώνα, να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ε, οι δεξιότητες μπορούν να προλάβουν τη φτώχεια. Οι δεξιότητες βοηθούν τους ανθρώπους να βάλουν πόντι στην αγορά εργασία. Και επίση, η πρόσβαση στην αγορά εργασία πρέπει να συνοδεύεται και με δίκαιες συνθήκες εργασίας ελάχιστη μισθή, καλή μισθή, που θα δίνει τη δυνατότητα καλού επίπεδου διαβίωση στους ανθρώπους. Πρόκειται και για την κοινωνική ε, προστασία. Η καλή κοινωνική προστασία υφίσταται όταν οι μη έχοντες μπορούν να επωφεληθούν και προσφέρει κανεί ωφέλη σε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ε, τα συνδυάσουν αυτά με πολύ καλά αναπτυγμένες υπηρεσίε. Αλλιώς όλα αυτά δεν λειτουργούν μακροπρόθεσμα. Για τη φτώχεια Κυρία Τρεμπέσιους, αν δει κανεί τη δυνατότητα των κρατών μελών να οργανώσουν την κοινωνική προστασία, πράγματι οι δυνατότητε δεν είναι ίδιε παντού σε όλα τα κράτη-μέλη, άλλο το επίπεδο κίνηση. Η Γερμανία μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από τη Ρουμανία. Όμω όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν κάτι. Και γι' αυτό και εμεί το υπογραμμίσαμε αυτό ε, στι συστάσει μα ανά χώρα. Και γι' αυτό είναι ακριβώ το λόγο όταν μιλάμε για την σύγκληση, προς τα πάνω βέβαια, λέμε θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι διαφορετικές ε, συνθήκες στα κράτη-μέλη. Δεν πρέπει να είμαστε τυφλοί, να έχουμε τα πόδια στη γη, ε, να ξέρουμε βέβαια ότι όλοι μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα. Χρειαζόμαστε σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στην Ευρωζώνη, αλλά και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Στα 27. Ο κοινωνικός πυλώνας θα βοηθήσει τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών να επιτύχουν τους στόχους τους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Και τώρα δίνω το λόγο στην ε, συνάδελφό μου την κυρία Ολσπόκ. Και συνεχίζουμε με τις ερωτήσεις για 1,5 λεπτό στον κύριο Παπαδημούλη. Παρακαλώ κύριε Παπαδημούλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα μιλήσω στα ελληνικά. Για μια ακόμη φορά θέλω να σας θέσω ένα θέμα που αφορά στην Ελλάδα, τη χώρα μου. Η Ελλάδα εξαιρείται των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αλλά έχει τεθεί ένας κοινός στόχος και από την Ελλάδα και από τους δανειστές από τον Αύγουστο του 2018 και μετά να μην χρειαζόμαστε μνημόνια και συναφείς δανειακές δεσμεύσεις, και να μπορούμε, όπως όλες οι χώρες κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, να δανειζόμαστε με λογικά επιτόκια από τις αγορές. Σήμερα μας ανακοινώσατε, κύριε Επίτροπε, ένα θετικό νέο, ότι η Κομισιόν αποφάσισε να βγει η Ελλάδα από τη διαδικασία περί υπερβολικού ελλείμματος με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αλλά εκκρεμεί και η απόφαση του Eurogroup για την αποσαφήνιση των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάψης του χρέους, που θα εφαρμοστούν μεν μετά το τέλος του προγράμματος, αλλά έχει συμφωνηθεί να προσδιοριστούν τώρα, για να υπάρχει ένας καθαρός οδικός χάρτης και για τους επενδυτές, και για τους Έλληνες, και για τις αγορές, και για, για όλα τα κράτη-μέλη, που θα βοηθήσει την Ελλάδα στην ανάκαμψη. Σας ρωτώ λοιπόν τι προτείνει, τι περιμένει, τι προσπαθεί η Κομισιόν εν ώψη του Eurogroup στις 15 Ιουνίου, προκειμένου να υπάρξει αυτή η συμφωνία η συνολική, από τη στιγμή που οι Έλληνες έκαναν πράξη τις δεσμεύσεις τους. Και το δεύτερο, δώστε μας λίγο παραπάνω στοιχεία για το πώς ήταν το δημόσιο έλλειμμα στην Ελλάδα το 2015 το 2016, ποιες είναι οι προβλέψεις το 2017 και τι θα σημάνει πρακτικά η έξοδος της Ελλάδας από τη διαδικασία περί υπερβολικού έλλειμματος. Thank you. Ε, ε, I can't see that she is here. Ε, κυρία Κούνεβα. Δεν ξέρω αν είναι εδώ. Δεν θα χρησιμοποιήσω το χρόνο, θα το δώσω στην ε, ε Κομισιό για να απαντήσει. Ερνέστο να έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτα, ε, οι συγκεκριμένες συστάσεις για την Ισπανία. Όσον αφορά στην πάταξη της διαφθοράς, ε, είναι καλοδεχούμενες οι προτάσεις, είναι πολύ συγκεκριμένες. Έχω όμως δύο ζητήματα. Πώς θα διασφαλίσει η Κομισιόν ότι θα εφαρμοστούν και δεύτερον υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με τις δημόσιες συμβάσεις για τα δημόσια έργα. Αυτά σχετίζονται με τα δημόσια οικονομικά και τη διαφθορά. Έχετε συζητήσει αυτό το θέμα με τις Ισπανικές Αρχές. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δεύτερο ερώτημα, περνάω στη σύσταση για τη Γερμανία. Ήδη αναφέρατε ότι υπάρχει πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαχών το θέμα όμως ε, είναι ότι δεν έχετε ακόμα κηρύξει διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών και με ορθρωτικές δράσεις. Πόσο μεγάλο πρέπει να είναι λοιπόν το πλεόνασμα και για πόσο καιρό πρέπει να διαρκεί πριν το κάνετε, γιατί είναι νομίζω στις αρμοδιότητές σας και είναι μία από τις μεγαλύτερες ανισορροπίες που έχουμε στην ε, Ευρωζώνη. Και υπάρχει και μια τρίτη ερώτηση για τον Επίτροπο Μοσχοβιστή. Είπατε ότι στον Ευρωζώνη έχουμε πολύ μικρή ζήτηση, ένα αρνητικό χάσμα παρά την ανάκαμψη και την ευελιξία που έχει δώσει η Κομισιόν. Συμφωνείτε με αυτό που είπε χθε ο κύριος Ντράγκη ότι η Ευρωζώνη χρειάζεται μια δημοσιονομική δυνατότητα με δανειοληπτική ικανότητα δανειοδοτική ικανότητα έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτό που είχαμε στο παρελθόν, μία διπλή ύφεση και επίσης σε επίπεδο ΑΕΠ πόσο μεγάλη πρέπει να είναι αυτή η ικανότητα και τι νομίζετε ότι θα αλλάξει με όλα αυτά. Ευχαριστώ. Τζιν Λάμπερτ ε, είναι η επόμενη ομιλήτρια, δεν την βλέπω. Πήρα 30 δευτερόλεπτα από το χρόνο της. Ναι, όντως.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 Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ και τους επιτρόπους. Ε, θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι, βρίσκομαι σε σύγχυση λιγάκι, γιατί μιλάμε εδώ για μέτρα τα οποία θα έπρεπε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, αλλά η πραγματικότητα που λέτε ότι γνωρίζετε ή γιατί έρχεστε σε επαφή με τα κρατημέλη, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ε, στην Ευρώπη υπάρχουν πάνω από 120 εκατομμύρια φτώχοι και αυτή είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόσετε και συνεχίζετε να εφαρμόζετε προσπαθώντας να δικαιολογήσετε το δικαιολόγητο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προτείνεται και επιβάλλετε στα κράτη-μέλη έχουν οδηγήσει σε κοινωνική σφαγή. Αλλά εσείς συνεχίζετε ε, ατάραχοι χωρίς να ομολογείτε ότι αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, ένα δικαιολόγητο λάθος το οποίο σήμερα όχι μόνο καθορίζει τη ζωή των 120 εκατομμυρίων φτωχών στην Ευρώπη αλλά θα και στη θυσία των μελλοντικών ε, γενεών και αυτό στο όνομα ποιου, ποια αξία, ποιο είναι ο στόχο που πρέπει να επιτύχουμε. Γιατί δεν θα πρέπει κανεί ε, να εφησυχάζει όταν τα κράτη-μέλη τα καταφέρνουν με τι παράλογε παραμέτρου που επιβάλλεται. Γιατί αυτά που μα επιβάλλεται αυτή τη στιγμή οδηγούν στην απόλυτη φτώχεια, οδηγούν στην φτώχεια στο σύνολο τη Υπήρου. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι χαρακτηριστική. Συνεχίζουμε να οδηγούμε σε λιμοκτονία ένα λαό, εφαρμόζουμε μέτρα τα οποία όμως δεν δημιουργούν απασχόληση, μέτρα τα οποία δεν επιτρέπουν σε κάποιους να φύγουν από τη φτώχεια και να ξαναμπούν στο χώρο της εργασίας. Καταστρέψατε λοιπόν όλα εκείνα τα οποία Ακόμα και αν εφαρμόζονταν μέτρα σήμερα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρουν ενδιαφερόμενη θέση απασχόλησης. Και πότε επιτέλους ε, θα αποφασίσετε, γιατί είναι η μόνη ερώτηση που κάνω, πότε θα αποφασίσετε και θα συνειδητοποιήσετε ότι έχετε κάνει τεράστιο ατόπιμα, μεγάλο λάθος στην πολιτική που εφαρμόσετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τον ε, κύριο Επίτροπο ε, θέλω να πω ότι όσον αφορά τις στάσεις αναχώρα, καλές είναι και σωστές οι προτάσεις, ανάπτυξη και όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως ε, και θα πρέπει να υπάρχει μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, η οποία θα πρέπει να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Όμως, εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε όσον αφορά τις συστάσεις αναχώρα να είσαστε πιο συγκεκριμένοι και θα πρέπει να συμπεριλάβετε του κοινωνικού εταίρους. Γι' αυτό λοιπόν, όσον αφορά τη δική μου τη χώρα, την Αυστρία, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στι δικέ μα συστάσεις ανά χώρα. Η Κομισιόν λέει ότι θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν ε, οι συντάξει. το σύστημα τη υγεία και το σύστημα τη παιδείας. Αν τα δει κανεί επιφανειακά, σωστά τα λέει. Μόνο που, όπω συχνά συμβαίνει, η λεπτομέρεια είναι εκείνη που καθαρίζει τι εξελίξει. Και θέλω να σα πω ότι στην Αυστρία πράγματι αυξάνονται οι δαπάνες για τις συντάξεις, μακροπρόθεσμα όμως θα μειωθούν οι δαπάνες και οι ε, ηλικίε συνταξιοδότηση των 65 ετών ίσως να είναι χαμηλό αυτό το όριο, αλλά ξέρετε στην Αυστρία εμεί έχουμε πάρα πολλέ πρόορε συνταξιοδοτήσει. Αυτέ λοιπόν οι πρόορε συνταξιοδοτήσει οδηγούν στο να μην μπορούν να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις. Στο σύστημα υγεία. πράγματι εκεί αποδίδεται τεράστια σημασία και προβάλλονται ιδιαίτερα τα νοσοκομεία, Όμω, εκεί που μιλάτε για τη φορολογική πολιτική δεν είναι σωστό να λέτε ότι θα πρέπει πρέπει να αυξηθούν οι φόροι στην ενέργεια. 15% επιβάλλεται ο φόρο στην ενέργεια και θα ήταν αντιπαραγωγικό να αυξηθεί περαιτέρω η φορολόγηση ενέργεια στην Αυστρία. Κι εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Μοσκοβισή ότι υπάρχει, υπάρχει πράγματι τεράστιο πρόβλημα ζήτησης. Άρα δηλαδή ίσως θα έπρεπε να αλλάξει η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί από ό,τι φαίνεται με αυτό το σύστημα δεν υπάρχει όθηση στη ζήτηση και εξάλλου οι νομισματικές πολιτικές αυτές που εφαρμόζονται, οι πολιτικές αυτές είναι υπερβολικές. Δεν επιτρέπουν την πραγματική ανάκαμψη. Αν δούμε λιγάκι το τι συμβαίνει στη Γερμανία και στην Ολλανδία, ε, αυτό το υπερβολικό πλεόνασμα αυξήθηκε περαιτέρω. Μία συγκεκριμένη τώρα ερώτηση. Υποτίθεται είμαστε σε μια νομισματική ένωση. Υπάρχουν όμως παρόλα αυτά οι ανισορροπίες. Και αντί λοιπόν να επιβάλλεται συγκεκριμένη πολιτική επενδύσεων σε χώρες που έχουν ένα υπερβολικό πλεόνασμα, γιατί δεν κάνετε αυτό που γινόταν πάντα σε μια πραγματική νομισματική ένωση. Δηλαδή, αυτοί που έχουν πλεόνασμα να ενισχύσουν εκείνους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε υπερβολικό έλλειμμα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο, το οποίο έχει άμεσα σχέση με την εφαρμοζόμενη πολιτική. Εγώ το βάζω αυτό το θέμα στο τραπέζι, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάκαμψη ε, και αυτό αφορά προφανώς την νομισματική ένωση στην οποία αναφέρεστε κι εσείς. Δηλαδή, Ερωτώ, γιατί το πλεόνασμα, το υπερβολικό, να μην συνδεθεί άμεσα με το υπερβολικό έλλειμμα. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ευχαριστώ, Ντομινίκ Μαρτά. Δεν είναι εδώ. Και τώρα... Δεν βλέπω τον κύριο Μαρτά, αν περιπτώσει. Ε... να περάσουμε τώρα στους επιτρόπους. Πρώτα ο κύριος Ντομπρόφσκης, παρακαλώ. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Τέθηκαν μια σειρά από ερωτήματα. Για τις συστάσεις αναχώρα και την Ισπανία πιο συγκεκριμένα, την ε, ερώτηση 1, στη σύσταση μάλλον υπαρθμών 1, αναφερόμαστε και στην ανάγκη να ενισχυθεί το πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και συστήνουμε στην Ισπανία να δημιουργήσει ένα ε, σύστημα ενίσχυσης εθνικό ε, των δημοσίων συμβάσεων που να καλύπτει όλα τα επίπεδα. Για να επανέλθω τώρα στο θέμα του γερμανικού πλεονάσματος. Ξεπερνάει τις τιμές αναφοράς και ε, αυτό γίνεται για δεύτερη τρίτη φορά οπότε γι' αυτό η Γερμανία είναι στην κατηγορία αυτή ε, της διαδικασίας περί μακροοικονομικής αστάθειας, ανισορροπίας. Αλλά δεν θεωρούμε ότι αυτό θα συνεχιστεί με βάση τα στοιχεία που έχουμε και για τους μισθούς. Οπότε δεν θεωρούμε ότι πρέπει να πάμε προς τη διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών. Ακόμα. Τώρα, για την ε, δημοσιονομική δυνατότητα της Ευρωζώνης. Αυτό τώρα ε, προκαταλαμβάνει κάπως ε, το έγγραφο για την Οικονομική Ένωση που θα υποβληθεί αύριο, οπότε δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό. Πάντως αναπτύσσουμε αυτή την έννοια με βάση αυτά τα οποία αναφέρονται στην έκθεσή μας για να μπορέσει να λειτουργήσει ε, αυτή η προσπάθεια σταθεροποίησης ε, της Ευρωζώνης. Αλλά θα παρουσιάσουμε το έγγραφο αυτό αύριο. Για τα ερωτήματα τώρα που τέθηκαν ε, για την Αυστρία πιο συγκεκριμένα για την πρόορη εξεδότηση Στην Αυστρία, μεταξύ των συστάσεων, μιλάμε για τη βιωσιμότητα των στεξιωτικών συστημάτων και η αντιμετώπιση της ε, διευρυμένης προσδεξιδότησης είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό. Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας ε, και τη συμμετοχή των γυναικών, των ανθρώπων που προέρχονται από τη μετανάστευση ε, υπάρχουν σχετικέ συστάσει, όμω το θέμα τη πρώτη ταξιδιώτηση ε, σχετίζεται με τη βιωσιμότητα του ταξιδιωτικού, του συστήματο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Τάισεν. Uh, κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αυτές που έχουν να κάνουν με τις ε, κοινωνικές πτυχές ήδη έχουν απαντηθεί από τον Αντιπρόεδρο, νομίζω, κύριο κύριος Euh, euh. Τρεις συμπληρωματικές απαντήσεις. πρώτη για την Ελλάδα. Να εξηγήσω γιατί ε, παρόλο που υπήρχαν οι απαιτήσει δεν προχωρήσαμε στην Ελλάδα ε, να, γίνει άρση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Όντως ε, υπάρχουν τα νούμερα, δεν τα έχω ακριβώς αυτή τη στιγμή, όμως έχουμε πέσει αρκετά κάτω. Οι προσπάθειες ε, σε επίπεδο ε, πρωτογενούς ελλείμματος έχουν πέσει, ε, έχουν αποδώσει αρκετά, τα 4,2% το 2017, 3,7% είναι πάνω από τον στόχο δηλαδή που είχαμε θέσει αρκετά, αρχικά. Φυσικά αυτή η καλή απόδοση θα συνεχίσει και του χρόνου και αυτά είναι καλά νέα και όπως ξέρετε οι συζητήσεις για τη δεύτερη αξιολόγηση συνεχίζονται σχετικά με το δημοσιονομικό δρόμο που θα ακολουθήσει η Ελλάδα και θα ξανασυζητηθεί στο Eurogroup στις 15 Ιουνίου. Στην περασμένη συνάντηση είχαμε σημαντική πρόοδο, όπως το ξέρετε, άλλωστε, όμως δεν μπορέσαμε να φτάσουμε σε καταληκτικό συμπέρασμα. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει στο επόμενο Eurogroup. Η Κομισιόν όπως πάντα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παίξει ένα ρόλο ως ε, ειλικρινής διαμεσολαβητής. Εγώ συμβουλεύω τις ελληνικές αρχές ε, να αναλάβουν και αυτές τις δικές τους ευθύνες. Όταν κοιτάζω τα προαπαιτούμενα, τα οποία είναι πάρα πολλά, 140 αν δεν κάνω λάθος, ε, και είναι και πολύ φιλόδοξα, εντάξει, ξεκάθαρα βρίσκομαστε στο σωστό δρόμο. Ξέρω όμως επίσης ότι υπάρχουν και κάποιες απαιτήσει που πρέπει να εκπληρωθούν πριν επιληθεί το θέμα του χρέους. Ελπίζω ότι και αυτά ε, θα τα επιλύσουμε με λογικό τρόπο τις επόμενες εβδομάδες. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η Κομισιόν περιμένει αυτή την γενικότερη συζήτηση για να επανέλθει ε, το θέμα. Η διαδικασία για το υπερβολικό έλλειμμα για την Ελλάδα θα έχει κάποιο νόημα αν έχουμε συμφωνία. Όπως και να έχει θα έχει κάποιο νόημα, αλλά αν έχουμε και τη συμφωνία ακόμα καλύτερα. Και ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε συμφωνία. Τα ερώτηματα τώρα που τέθηκαν για την Αυστρία. Το 2013 13,9% του ΑΕΠ ήταν ε, οι δαπάνες ε, για τις συνταξίες ε, θα μειωθεί κατά 0,5% μέχρι στο επόμενο διάστημα που είναι πολύ παραπάνω από το 0,3% μείωση που περιμέναμε. Είναι μεγάλο θέμα, ε, μεγάλο επίτευγμα και σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού ε, συστήματος στην Αυστρία αύξησε την ηλικία ε, συνταξιοδότησης, όμως υπάρχει αύξηση στις συνταξιοδοτικές δαπάνες και ακόμα δεν έχει οριστεί ε, το πώς θα σταθεροποιηθεί το ζήτημα αυτό. Κατά την άποψη της ε, ε, Κομισιόν πρέπει να υπάρχει ας πούμε μια αυτόματη ρύθμιση που θα βασίζεται στο προσδόκιμο διαβίωσης. Δεν θα επανέλθω σε αυτό. Θα περάσω στο τρίτο σημείο που αναφέρεται στην έλλειψη ζήτησης επαναλαμβάνω με αυτόν τον τρόπο τις σκέψεις μου σχετικά με τις επενδύσεις και την ανάγκη για μια δημοσιονομική ικανότητα. Θεωρώ προσωπικά όντως ότι η πρόταση του κυρίου Ντράγκη πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να σημαίνει ε, ότι σε τέσσερα χρόνια από τώρα θα συνεχίσουμε να συμφωνούμε. Ένα Άλλο θέμα που έχει να κάνει με τη Γερμανία και την Ολλανδία είναι η αύξηση των μισθών. Δεν εξαρτάται από μας να πιλωτάρουμε την πολιτική οποιασδήποτε χώρας. Εμείς κάνουμε κάποιες προτάσεις γιατί θεωρούμε ότι με τη σύστασή μας ε, αυτή ε, δίνουμε μια πολύ συγκεκριμένη και σχετική απάντηση στο ζήτημα. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο Catch the Eye. Ο κύριος Μπούλμαν έχει το λόγο. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα από τον κύριο Ντομπρόφσκη. Και κύριο Ντομπρόφσκης... Ε, ακούστε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι και οι τρει σα, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, ε, προσπαθείτε για περισσότερη και καλύτερη σύγκληση. Και πρέπει να σα υποστηρίξουμε προ την κατεύθυνση αυτή Χρειάζεται, το είπε ο κ. Χόκμαρκ, πρέπει να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση, πρέπει να πάμε προ την κατεύθυνση αυτή. Όμω υπάρχουν ακόμα χώρε που έχουν επιμέρου προβλήματα, έχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Κάποιε άλλε χώρε έχουν μεγαλύτερο περιθώριο. Αναφέρετε στην έκθεσή σα αυτό. Τέθηκε το ερώτημα από του συναδέλφου ε, τι θα γίνει με τι χώρε τι πλεονοσματικέ. Ιδιαίτερα σε μία χώρα ε, πόσο μεγάλο πρέπει να είναι πια το πλεόνασμα για να κάνει κάτι Κομισιόν γι' αυτό και δεν απαντήσατε στο ερώτημα αυτό απευθείας. Είπατε δεν αναμένω ότι θα αυξηθεί κι άλλο, αλλά θέλω να επανέλθω. Γίνεται ένας διάλογος εδώ, έτσι. Ένας επικοδομητικός διάλογος μαζί μας. Φαντάζομαι ότι θα έχετε διάλογο και με άλλες χώρες. Τι λένε με οι χώρες. Οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, τι λένε όταν τους λέτε εσείς. Σας παρακαλώ χρησιμοποιήστε το περιθώριο λιγμών που έχετε για να ενισχύσετε την προσπάθεια που κάνουμε για μεγαλύτερη σύγκληση. Ποια είναι η αντίδραση στις χώρες αυτές. Εμείς θα θέλαμε να γνωρίζουμε ως ευρωβουλευτές πού έχει φτάσει ο διάλογος αυτός. Ξέρω ότι για το, το six-pack ήταν πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο ε, πλευρές στην ανισορροπία. Ευχαριστώ, ο Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα ερώτημα προς τον Επίτροπο Μοσκοβισή για την χώρα μου, την Πορτογαλία. Αναφερθήκατε στο πολύ καλό νέο ότι η Πορτογαλία θα εγκαταλείψει την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Και αυτό βεβαίως δεν βασίζεται μόνο στην μείωση του ελλείμματος, αλλά βασίζεται και σε μια γενικότερη οικονομική βελτίωση. Εδώ και ε, τρία τρίμηνα είμαστε σε ρυθμού ανάπτυξη πάνω από το μέσο όρο τη Ευρωζώνη. Υπάρχει βελτίωση στην απασχόληση, υπάρχει μια σταθεροποίηση του χρηματοοικονομικού συστήματο. Λαμβάνοντα υπόψη όλα αυτά τα θετικά στοιχεία, πιστεύετε ότι θα έχουμε και καλά νέα σε ό,τι αφορά του οίκου αξιολόγηση για το χρέο τη Πορτογαλίας και την αξιολόγησή του. θα υπάρξει ένα πιο θετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα επιτρέψει την Πορτογαλία και σε άλλες χώρες να αντιμετωπίσουν καλύτερα το θέμα των ε, κόκκινων δανείων. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Σούλτσε, παρακαλώ, έχει το λόγο. Δεν θέλετε ερώτηση. Η κυρία Σατιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους επιτρόπους. Ε, μας ε, ζωγραφίσατε μια εικόνα η οποία δείχνει βελτίωση, αλλά είμαστε ακόμα ευάλωτοι. Ο καλύτερος τρόπος να πατάξουμε την φτώχεια είναι να έχουμε ε, επαγγελματική ολοκλήρωση. Υπάρχουν τρεις μοχλοί για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό. Πρώτον, τα 10 επαγγέλματα που ε, έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση σήμερα δεν υπήρχαν πριν από 10 χρόνια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πως η κατάρτιση ε, μέσω πτυχίων στην ουσία ε, δεν ταιριάζει πια στην δυνατότητα αντίδρασης που πρέπει να έχουμε στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την κατάρτιση ε, και να μπορέσουμε να έχουμε δεξιότητες οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλα τα κράτη-μέλη. Αλλιώς ε, θα έχουμε πολύ, ε, πολλές προσπάθειες οι οποίες θα είναι χωρίς αποτέλεσμα. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι δεξιότητες να αποτελέσουν κομμάτι των συστάσεων αναχώρα. Δεύτερον, Έχετε δείκτες σχετικά με την φυγή εγκεφάλων από την Ευρώπη προς ε, τρίτες χώρες ε, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ώστε αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στην Ευρώπη. Η καινοτομία και η έρευνα είναι ένα θέμα, αλλά το να κρατήσουμε και τους ανθρώπους αυτούς εδώ είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Τρίτον, ενίσχυση της κινητικότητας ε, στις ευρωπαϊκές ε, χώρες. Νομίζω ότι αυτό είναι μια σύσταση που πρέπει να γίνει στο εσωτερικό των κρατών μελών, ε, στα 27 κράτη-μέλη, γιατί και η κινητικότητα είναι μια αγγίση για την πάταξη της ανεργίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυρίδης, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρατήρηση από τη συνάδελφό μου, παρόλο που δεν ήταν αυτός ο λόγος που θα ρωτούσα. Labor mobility είναι ένα πράγμα, αλλά brain drain είναι άλλο πράγμα και εμείς οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, ειδικά Κύπρος, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία και πολλές άλλες, υποφέρουμε γιατί the best of the best εγκαταλείπουν τις χώρες μας και μετά φεύγουν για άλλες χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως έρχομαι στο ερωτήματα μου, θα είναι δύο. Το ένα γενικό, το άλλο ειδικό. Το γενικό είναι το εξής. Πριν μερικούς μήνες είχαμε εδώ στο Econ Committee συζήτηση με τον επικεφαλής του Eurogroup. Σας ανησυχεί κύριε Επίτροπη το γεγονός ότι πριν μερικούς μήνες χωρίς να αλλάξει οτιδήποτε στο τραπέζι εδώ κουβεντιάζαμε για διορθωτικά μέτρα για εκείνες τις χώρες οι οποίες είχαν excessive imbalances. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή η αντιφατικότητα στη διαδικασία σας ανησυχεί. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι about social matters, Madam Tyson. Τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κατά 21% έχουν δεσμευτεί για την Κύπρο για θέματα προσβασιμότητας των μειονεκτουσών ομάδων, όπως αναπήρω. Και καλά έγινε. Σας μεταφέρω όμως ακόμα ένα πρόβλημα. Οικογένειες με παιδιά τα οποία έχουν νοητική στέρηση, όταν γίνουν 21 χρονών, δεν έχουν πουθενά να τα αφήσουν για φροντίδα και καταλήγουν είτε στα ψυχιατρία, είτε σε γυροκομεία. Έχετε κάτι να μας πείτε. Ε, Ευχαριστώ. Η Χέλγα Stevens δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ κυρία Τάισεν. Το Βέλγιο δεν ε, έχει μια πολύ καλή θέση στην δική σας έκθεση, αλλά αυτό δεν μας εκπλήσει, αν κανείς σας ξέρει. Μόλις ξεφύγαμε από την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, Έχουμε ιδιαίτερα υψηλό χρέος και έναν ε, προϋπολογισμό που ούτως ή άλλως ε, δεν είναι κελισμένος. 1,7 δις ε, μας λείπουν πρέπει να ανακαινήσουμε, να ανανεώσουμε τους πυρηνικούς σταθμούς ενέργειας. Έχουμε ένα πολύ κακό φορολογικό σύστημα και μέχρι το 2014 όλα τα πολιτικά κόμματα ε, είχαν ε, κατά νου και ήταν ξεκάθαρο ότι χρειαζόμασταν μία εθνική μεταρρύθμιση. Η διχοτομία αυτή η διαφορά μεταξύ των δύο μερών στο Βέλγιο πρέπει να επιληθεί με μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις. Γιατί λοιπόν η Κομισιόν δεν αναφέρεται σε αυτό το ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα. Τελευταία ερώτηση. Την κυρία Ρούχανεν. Ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε. Η Φιλανδία υπήρξε μοντέλο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει όντως στηρίσει όλους τους κανόνες ε, και στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και σε κάθε άλλο επίπεδο. Όμως έχουμε μηδενική ανάπτυξη. Η μακροχρόνια ανεργία αυξάνεται δομές ε, της, ε, του κοινωνικού κράτους ε, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τι συμβαίνει λοιπόν με τη Φιλανδία. ποιο είναι το πρόβλημα. Η Σουηδία κατάφερε να ξεφύγει γρήγορα από την κρίση και τα πάει πολύ καλά. Η μόνη ξεκάθαρη διαφορά που έχουμε με τη Σουηδία είναι ότι η Σουηδία δεν είναι ε, μέρος του ευρώ. Δεν μας κάνει καχύποπτους αυτό. Ίσως το ευρώ να ευθύνεται για όλα αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ε, όλες λοιπόν οι ερωτήσεις θα κάνεις ε, τέθησαν. Ε, ως εκ τούτου, κύριε Ντομπρόφσκι, ξεκινάμε με εσά και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το θέμα του ε, πλεονάσματος ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ε, δεν συμφωνώ με αυτό που ελέγχθη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει απολύτως τίποτα. Δεν είναι αλήθεια. Και ε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Γερμανία έβαλε την, η Επιτροπή έβαλε τη Γερμανία σε αυτή τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών με τον ε, συνοδεύοντα μηχανισμό εποπτείας. Και αυτός είναι και ο λόγος γιατί σε αυτή τη διαδικασία η αξιολόγησή μας είναι ότι υπάρχουν ανισορροπίες, όχι βέβαια υπερβολικές. Κατόπιν, ετέθη το ερώτημα ποια είναι τα επιχειρήματα που προβάλλει η Γερμανία αλλά και η Ολλανδία για το ίδιο ακριβώς θέμα. Πρώτα απ' όλα, να σας πω ότι ακούμε ότι και οι δύο χώρες ε, έχουν την πούληση να αυξήσουν τις ε, δημόσιες επενδύσεις και πράγματι διαπιστώνεται κάποια πρόοδος στην ε, πραγματοποίηση δημόσιων επενδύσεων στη Γερμανία. Λήφθησαν μία σειρά πρωτοβουλειών προς αυτή την κατεύθυνση. Κατόπιν υπάρχουν και κάποια επιχειρήματα που αφορούν στη μέθοδο. Η Γερμανία ισχυρίζεται ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσει κανείς ε, το πλεόνασμα σε σχέση με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πλεόνασμα σε σχέση με τρίτες χώρες. Η Γερμανία, αν ε, περιόριζε τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες, θα βοηθούσε την ευρωπαϊκή οικονομία, ότι μαθηματικά ποτίθεται αυτό θα έλυνε το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που προβάλλει η Γερμανία και θα το αξιολογήσουμε. Τώρα, στην περίπτωση της Ολλανδίας είναι ότι γίνεται επανεξαγωγή σε χώρες Ευρωζώνης λόγω των εισαγωγών που γίνεται, γίνονται από το Ρότερνταμ. Αυτό το επιχείρημα προβάλλουν, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να εισακουστούν τα δικά μας τα επιχειρήματα, να υπάρχει βούληση να αυξηθούν οι δημόσιες επενδύσεις στην Ολλανδία. Η κυρία Τάισεν. Κυρία Πρόεδρε. Για τις επενδύσεις ε, στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την ενίσχυση της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου φυσικά κάναμε περισσότερα φέτος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η κυρία Μόρεν Σαρτιέ το ανέπτυξε Πολύ σωστά και γι' αυτό το βάλαμε και στον πυλώνα 1 των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αν δούμε τις διαφορετικές στατιστικές, ε, αν δείτε ποιοι είναι στην ανέχεια, ποιοι είναι άνεργοι, θα δείτε ότι οι δεξιότητες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Η ανταγωνιστικότητα, η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας χρειάζεται όχι μόνο ανθρώπους με ταλέντο, αλλά και ανθρώπους που θα έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να χρησιμοποιήσουν το δυναμικό που έχουν στην αγορά εργασίας και να αναπτύξουν με αυτόν τον τρόπο όλη την κοινωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό ε, πρέπει να παραμείνει ε, στην κορυφή της ε, των προτεραιοτήτων της Κομισιόν. Γι' αυτό φτιάξαμε και αυτή την ατζέντα για τις δεξιότητες που δημοσιοποιήσαμε πριν από μερικούς μήνες. Όπως σας είπα ήδη, πρέπει να δούμε το θέμα της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων. στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτό καλύτερα, πώς θα βοηθήσουμε τον κόσμο να ε, διαμορφώσει τις δεξιότητές του έτσι ώστε να έχει καλύτερη αναγνώριση σε τυπικό επίπεδο ε, της άτυπης μάθησης ε, των άτυπων δεξιοτήτων που κατέχει. Επίσης, η φυγή εγκεφάλων, το brain drain, είναι ένα πολύ γνωστό πρόβλημα κινήσεις εκτός Ευρώπης αλλά και εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυξάνονται. Για κάποια κράτη-μέλη το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Βλέπουν ε, πολλά άτομα να φεύγουν από τη χώρα. Και το πρόβλημα αυτό, όπως σας ανέφερα ήδη, το έχουμε αναγνωρίσει, περιλαμβάνεται στην ατζέντα για τις δεξιότητες και στην ουσία αποτελεί ε, αυτό η ατζέντα έναν τρόπο να βρούμε τις βέλτιστες πρακτικές ε, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το brain drain και αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Για το θέμα των ατόμων με αναπηρία. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και όλα τα κράτη-μέλη της ξεχωριστά, έχουν υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ένα από τα στοιχεία αυτής της σύμβασης ακριβώς αναφέρεται στο να μην ιδρυματοποιούνται τα άτομα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι γενικά είμαστε υπέρ ε, αυτών των υπηρεσιών που θα τους κρατήσουν έξω από τα ιδρύματα, που θα τους κρατήσουν στην οικογένειά τους ε, για να μην χρειάζεται να ιδρυματοποιηθούν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Μουσκοβίση, έχει το λόγο. Ένα ερώτημα μόνο μου τέθηκε και θα απαντήσω ε, για την Πορτογαλία. Είναι σαφές ότι η έξοδος από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος έχει να επιβραβεύσει σημαντικές προσπάθειες που έχει καταβάλει η χώρα αυτή. Όχι μόνο είμαστε πολύ κάτω από το 3%, αλλά είναι πλέον και κάτω από το 2%. Οπότε είναι ένα πολύ καλό νέο το οποίο καλωσορίζω εκ νέου και ε, επαναλαμβάνω επιβραβεύει τι προσπάθειε. Λέτε τώρα για του οίκου αξιολόγηση. Ε, δεν μπορεί η Κομισιόν να μιλήσει στου οίκου αξιολόγηση. Δεν το κάνουμε αυτό εμεί. Δεν έχει αλλάξει ο βαθμός της Πορτογαλίας, αλλά υπάρχουν, υπάρχει θετικό πρόσημο, θετικό προσανατολισμός. Ε, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να πω αυτό που είπα εδώ, είπα και σε πορτογαλικά μέσα. Από τη στιγμή που υπάρχει μια μακροοικονομική κατάσταση που βελτιώνεται, ε, από τη στιγμή που τα δημόσια οικονομικά είναι ε, βεβαίω πιο σταθεροποιημένα, παρότι υπάρχουν συστήματα χρέου, έτσι, μην το ξεχνάμε, ε, λογικό θα ήταν αυτοί που αξιολογούν την πορτογαλική οικονομία να αντιληφθούν ότι δεν μπορεί ο κίνδυνος ή το ρίσκο να το βλέπει κανείς σήμερα με τη ματιά του χθες. Είναι πολύ πιο λογικό να κάπως στην Πορτογαλία σήμερα από στο παρελθόν. Δεν μιλάω απευθεία στου οίκου αξιολόγηση, δεν μιλάμε μαζί του δηλαδή, αλλά μέσω αυτή τη απάντηση νομίζω ότι στέλνω ένα μήνυμα ε, και πρέπει να ειδωθεί θετικά ε, η εξέλιξη της πορτογαλικής οικονομίας η οποία ε, σίγουρα εμπνέει όλο και περισσότερη εμπιστοσύνη. Τέτοια και ένα ερώτημα για τη Φιλανδία και τη Σουηδία στο τέλο. Ακούστε, ο καθένα ε, έχει την άποψή του υπέρ κατά του ευρώ. Ε, αλλά καταρχήν η φιλανδική οικονομία δεν είναι σε τόσο κακή θέση. Υπάρχει και μια ευελιξία για τις διαστροτικές μεταρρυθμίσεις, ε, διότι πιστεύουμε ότι υπάρχει μια σαφής πολιτική ατζέντα. Το συζητήσαμε επί μακρόν με τον ε, Υπουργό όταν βλέπουμε την απόδοση των δημοσίων οικονομικών ε, είναι θετικά τα πράγματα. Τώρα, επειδή κάνετε αυτή τη σύγκριση με τη Σουηδία, δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το αν κάποιο είναι στην Ευρωζώνη ή εκτό. Η Σουηδική οικονομία όπως γνωρίζετε είναι πιο διαφοροποιημένη ε, πιο πολυσχηδής από εκεί πέρα η σουηδικη οικονομια οπως γνωριζετε ειναι πιο διαφοροποιημενη πιο πολυσχηδης απο εκει περα η καθε χωρα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα ατού της, τα πλεονεκτήματά της. Φαντάζομαι και οι Φιλανδοί φίλοι μας θα το πράξουν. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο πλάι της Φιλανδίας, όπως και όλων των χωρών της Ευρωζώνης, για να τις ενθαρρύνει, έτσι ώστε να κάνουν τις απαραίτητες ε, θετικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως τις ιδιαιτερότητες του καθένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μοσκοβισή. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, όλα τα μέλη ε, που έθεσαν τα ερωτήματα αυτά, ε, έξυπνα ερωτήματα, δύσκολα ερωτήματα. Οι επίτροποι προσπάθησαν να απαντήσουν, ε, στο μέτρο του δυνατού βέβαια. Θα επανέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση για να μπορέσουν να τεθούν ε, και άλλα ερωτήματα. Πάντως βλέπουμε ότι γίνονται βήματα προς τη κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.